Dear colleagues, dear Συνάδελφοι, φίλοι μου, μέλη των κοινοβουλίων, καλώς ξαναήρθατε. Δεν θα σταθώ για πολύ στην εισαγωγή, γιατί έχω κοντά μου ε, καταπληκτικές γυναίκες και πραγματικά εγώ η ίδια ε, πρέπει να εκφράσω το θαυμασμό μου. Έχω την ε, Λάμια Χατζή Μπασάρ που επιβίωσε από την ε, σεξουαλική σκλαβιά στο ΝΤΑΕΣ, στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Είστε από την ε, ομάδα πληθυσμού των Γιαζιντή. Είναι Είμαστε πολλοί εμείς ε, που δακρύσαμε στην Ολομέλεια τον περασμένο Νοέμβριο όταν λάβατε το βραβείο Ζαχάροφ για το κουράγιο σας και την τόλμη σας. Είσαστε ακτιβίστρια και περασπίστε των δικαιωμάτων των Γιαζιντή και πραγματικά ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για να μας καταθέσετε την προσωπική σας μαρτυρία. Και επίσης να καλωσορίσω και την Χαουάουα, με συγχωρείτε για την πολύ κακή μου προφορά, την Χαουάουα Ιμπραχήμ. Είστε δικηγόρος ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νικήτρια του βραβείου Ζαχάροφ, είστε λάβει το βραβείο Ζαχάροφ το 2005, για την εκπληκτική σας αφοσίωση και την... Ε, προσπάθεια που έχετε κάνει στην ε, περιοχή σας και για την προσπάθεια που κάνατε να πέσει φως στην υπόθεση των κοριτσιών που απήχθησαν από το Μπόκο Χαράμ. Εδώ λοιπόν και εγώ και οι συνάδελφοί μου στο Κοινοβούλιο έχουμε στηρίξει την ε, παγκόσμια εκστρατεία σας. Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας που βρίσκεται και υπό τη δική σας αιγίδα και είναι μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας σήμερα. Πραγματικά ανυπομονούμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες σας. Προηγουμένως, πολύ σύντομα να πω ότι εγώ ίδια, ο πρόεδρο Ταγιάννη, ο επίτροπο Γιώροβα, ακούσατε πόσο όλοι είμαστε αφοσιωμένοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να ενώσουμε τι δυνάμει μα και να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Για να υλοποιηθεί πλήρω και να έρθει σε πλήρη ισχύ η σύμβαση του ΙΕ τη Κωνσταντινούπολη για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων ε, αυτή τη βία. Ε, έχουμε κοινά ψηφίσματα και εργαζόμαστε σε όλα τα κράτη-μέλη για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν όσα προβλέπει η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, να ξεκινήσει ένα επικοδομητικό διάλογο σε συνεργασία με το Συμβούλιο τη Ευρώπη, να αρθούν οποιοδήποτε επιφυλάξει και να υπάρξει μηδενική ανοχή κατά της ατιμορρησίας. Αυτή θέλουμε να είναι η ουσιαστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θέλουμε να κοιτάξουμε τις διασυνδέσεις που έχουν το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και τη οικονομική χειραφέτησής τους. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, ε, υποστήριξή μας και την ελεγγύη μας σε γυναίκες και κορίτσια που είναι θύματα βίας, ε, γυναίκες και κορίτσια που χάνουν τη ζωή τους στο σπίτι τους, στα σχολεία, κορίτσια που το σώμα τους, το πλήρωσαν, με το σώμα τους πλήρωσαν το ταξίδι τους από τον ΤΑΕΣ προς την Ευρώπη. Κορίτσια και γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, που Ξαναγκάζονται να παντρευτούν άντρε που δεν γνωρίζουν καν, που κάνουν παιδιά στα 12 και στα 13 του. Αυτό σημαίνει ότι οι ευκαιρίε του να πάνε στο σχολείο και να γνωρίσουν την οικονομική χειραφέτηση είναι κάτι που το ξεχνάνε για όλη τη ζωή. Μιλάμε για εκατομμύρια κορίτσια που κινδυνεύει η υγεία του επειδή ε, δέχτηκαν σεξουαλική βία με τον ένα τον άλλο τρόπο. Με τρομερές τραυματικές εμπειρίες και μετατραυματικές, με ψυχολογικές ε, πληγές. Εδώ θα σας πω τι έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε εγκρίνει μια οδηγία κατά της εμπορίας των γυναικών, ε, εμπορία, ε, ε, οδηγία συγγνώμη, για την προστασία των ε, θυμάτων, για την καταπολέμηση των δολοφονιών γυναικών και έχουμε ζητήσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγία για την ε, ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Βλέπω ότι κοντά μας από το Κοινοβούλιο της ε, Σερβίας ήρθε και η Γκορντάνα. Καλώ ήρθες, είσαι πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αντιπρόεδρο μάλλον του Κοινοβουλίου της Σερβίας και επίση εσύ συγγήτρια για το θέμα μας. Αύριο λοιπόν στην Ολομέλεια η Γκορντάνα θα συνοψίσει τα πορίσματα του δικού μα εργαστηρίου. Γιατί είναι η οικονομική χειραφέτηση σημαντική γιατί ε, πρέπει να περάσουμε από τον φαύλο ε, κύκλο στον ενάρωτο. Γιατί η οικονομική χειραφέτηση είναι τρόπος να ξεπεράσουμε την βία. Όταν ε, τρώει, όταν τρώει μια γυναίκα ξύλο από τον άντρα, τον σύζυγό της, τον σύντροφό της, πολλές φορές δεν μπορεί να φύγει γιατί η δάλος δεν θα μπορεί να τραφεί ή να θρέψει τα παιδιά της. Και δεν έχει και την οικονομική ανεξαρτησία για να κάνει ελεύθερες επιλογές και να αποφύγει τη βία. Αμέσως λοιπόν θέλω να σας δώσω το λόγο σε εσένα Λάμια. Παρακαλώ. Εγγραφείτε για τη συζήτηση. Υπάρχει εκεί ένα έγγραφο που πρέπει να το έχετε λάβει. Ελπίζω να έχουμε πολλή συμμετοχή και μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Ε, η εγγραφή αρχίζει τώρα. Παρακαλώ, παραδώστε το έγγραφο στην ε, ε, γραμματεία μας. Λάμια, έχεις το λόγο για 10 λεπτά. Θα μιλήσει αραβικά η Λάμια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ήθελα να σας ευχηθώ έναν καλό εορτασμό σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, ιδίως τις γυναίκες που βρίσκονται στα χέρια του ΝΤΑΕΣ. Είμαι από τους Γιαζεντή και βασανίστηκα Βασανίστηκα και βιάστηκα. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα ανήλικα κορίτσια σαν και που έχουν πέσει θύμα βιασμού. Ως τώρα, 300.000 κορίτσια και γυναίκες βρίσκονται ακόμη στα χέρια των δυνάμεων του ΝΤΑΕΣ, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και γνωρίζει όλος ο κόσμος τι κάνει τον ΝΤΑΕΣ σε αυτά τα κορίτσια και σε αυτές τις γυναίκες. Και ως τώρα ε, ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει. Οι γυναίκες αυτές, τα κορίτσια, τα παιδιά βρίσκονται στα χέρια του ΝΤΑΕΣ. Είναι όμοιροι Τις πουλάνε και τις αγοράζουν καθημερινά. Βασανίζονται καθημερινά, βιάζονται καθημερινά. Τα παιδιά επίσης. Παιδιά που είναι όμεροι του Ντάις. τα οποία υποφέρουν αυτά τα βασανιστήρια. Παιδιά που τα έχουν απαγάγει από τις μανάδες τους, τα έχουν υποχρεώσει να φέρουν όπλα, τους διδάσκουν το Κοράνι και δέχονται πλήση εγκεφάλου. Πριν από ένα μήνα μόλις, δύο παιδάκια για ζυμπή, δύο αδέρφια, έφτασαν από το Σιντζάρ. Είχαν ε, μεταμορφωθεί πλήρως. Τους είχαν κάνει πλήση εγκεφάλου και αυτοπυρπολήθηκαν στην μάχη της Μοσούλης. Το Νταές δεν είναι απειλή λοιπόν μόνο για μας, τους Γιαζιντή. Εάν δεν καταπολεμήσουμε την φιλοσοφία του Νταές και την πολιτική τους, θα καταστούν παγκόσμια απειλή. Οι γυναίκες και τα παιδιά που επιβιώνουν των δοκιμασιών, των βασανιστήριων αυτών που τους επιβάλλει τον ΤΑΕΣ, που ξεφεύγουν ε, από αυτούς τους καταβλισμούς του Κορδιστάν, ε, βρίσκονται σε συνθήκες ε, πραγματικά ολέθριες. Ζητάμε από τον κόσμο ολόκληρο να μην ξεχάσει ότι υπάρχουν παιδιά, κορίτσια και γυναίκες που βρίσκονται στα χέρια του ΤΑΕΣ κυρίως από τον πληθυσμό των Γιαζιντή. Δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Δεν είναι λίγες αυτές που αυτοκτόνησαν λόγω όσων πέρασαν. Και υπάρχουν γυναίκες και κορίτσια που ονειρεύονταν να τελειώσουν το σχολείο, να σπουδάσουν. Είχαν όνειρα είχαν ελπίδε και φιλοδοξίε. Και εγώ ήμουν έτσι. Ήμουν μαθήτρια και πήγαινα στο σχολείο. Ήθελα να τελειώσω το σχολείο, ήθελα να σπουδάσω μετά. Το ΝΤΑΕΣ όμως μου ε, έκοψε τα φτερά και δεν με άφησε να ζήσω κανένα από τα όνειρά μου και τις φιλοδοξίες μου. Αυτό λοιπόν που ζητάω είναι ο κόσμος να κινητοποιηθεί, να βοηθήσει, να βοηθήσει τις γυναίκες και τα παιδιά που ζουν ακόμα στους καταβλισμούς του Κουρδιστάν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση της Γερμανίας που ξεκίνησε το πρόγραμμα της, ε, του κρατηδίου της Βάδης Βουτεμπέργης, ε, υποδεχόμενο 500 ε, γυναίκες και κορίτσια στη Γερμανία, ώστε να υποφεληθούν από την ψυχολογική υποστήριξη και να επιστρέψουν ε, στις σπουδέ τους στο σχολείο ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ελπίζουμε και απευθύνουμε έκκληση προς ολόκληρο τον κόσμο να σκεφτούν πραγματικά τις γυναίκες, να ασχοληθούν πραγματικά με τις γυναίκες και τη μοίρα τους, την τύχη τους, διότι οι γυναίκες μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο, μπορούν να ψηφίσουν τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Λάμια. Και είμαι βεβαία ότι εκπροσωπώ όλους τους εδώ παρόντες και όσους μας ακούνε μάλιστα μέσω από το διαδίκτυο ότι δεν θα πέσει σε κοφεύοντα αυτιά η έκκλησή σου σήμερα την ημέρα των γυναικών. Και θα δώσω το λόγο τώρα στην Αουάια Ιμπραχήμ. Και πάλι σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κυρία Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι τέτοια μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Αλλά μια μας συγκίνησε σε όλους. Είσαι ζωντανό παράδειγμα θάρρους και αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη που είσαι εδώ. Καλή ημέρα των γυναικών, λοιπόν. Είχα ετοιμάσει μερικές παρατηρήσεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αλλά ε, όπως καθόμουν εδώ και έχω έρθει αρκετέ φορέ. με τιμήσατε με το βραβείο Ζαχάροφ το 2005. Σκέφτομαι λοιπόν σε αυτά τα χρόνια τι έχω κάνει διαφορετικό, τι περισσότερο μπορώ να πράξω. Τι έχετε κάνει εσεί. τι μπορείτε εσεί να πράξετε επιπλέον. Εορτάζουμε την ημέρα των γυναικών. Είχαμε καλές εξαίρετες ε, ομιλίες από τους προσκεκλημένους. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μιλήσω από καρδιάς, απευθυνόμενη στη δική σας την καρδιά. Τρία θέματα που ίσως να είναι και διαφιλονικούμενα, γιατί είναι κάποιες σκέψεις. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να, ακούσουμε, να μιλήσουμε και για αυτά που θέλετε εσείς να ακούσετε και όχι αυτά που θέλουμε εμείς να σας πούμε. Θα μιλήσω λοιπόν για τη γυναίκα και για την οικογένεια. Εορτάζουμε λοιπόν την ημέρα των γυναικών. Την πλατφόρμα του Πεκίνου, πλατφόρμα δράσης. Στόχους ανάπτυξης της χιλιτίας, στόχους αηφορίας που έχουμε ορίσει. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα σας κουράζουν αυτά. Ωραία. Ως μητέρες τι έχουμε κάνει, ως γυναίκες τι έχουμε κάνει και ως γυναίκες, ως αγωνίστριες, συναγωνίστριες τι μπορούμε να κάνουμε. Το 2014 το πέρασα προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι το Μποκοχαράμ και ποια είναι η σχέση τους με τα κορίτσια που έχουν απαγάγει. Το 2015 είχα την ευκαιρία στην Ιορδανία να αντιληφθώ λίγο τι είναι το η οργάνωση Ισλαμικό κράτος. Είπε η άλλη ότι είναι, η Λαμία ότι είναι αδελφή. 200 εκατομμύρια άνθρωποι και ένα κομμάτι της χώρας το έχει καταλάβει τώρα η Μποκοχαράμ. Τα νούμερα των απαγωγών ή της σεξουαλικής σκλαβιάς ε, είναι σχεδόν τίποτα μπροστά στα νούμερα αυτών που έχουν καταλάβει και υποδουλώσει. Μπορεί πρόσφατα να, να αντιμετώπισε ο τακτικός στρατός ε, το χαλιφάτο της μποκοχαραμα αλλά στον Ήγυρα, η γειτονική χώρα, όμορη χώρα, το Τσάτ, το Καμερούν, ακόμα έχουν έντονη παρασία. Είναι παρουσία. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την περιοχή και ελπίζω να ακούσετε εδώ από τις μαρτυρίες και οι βουλευτές για να αναλογιστείτε τι μπορείτε να κάνετε, τι δουλειά μπορείτε να προσφέρετε στους ανθρώπους που βρίσκονται και κυρίως τις μητέρες, τους γονείς και αυτό τον πλούτο, αυτά τα θύματα της Μποκοχαράμ, τα παιδιά της Μποκοχαράμ. Όλος ο μόχθος που κάνει ένα χωριό ολόκληρο στην Αφρική είναι να μεγαλώσει ένα παιδί. Το παιδί δεν ανήκει στον πατέρα ή στη μητέρα, αλλά σε ολόκληρο το χωριό. Τα κορίτσια αυτά που είναι τώρα δούλες, σεξουαλικές σκλάβες της Μποκοχαράμ, επιστρέφουν με παιδιά, με παιδιά, εκατοντάδες παιδιά. Γιατί ήταν χιλιάδες οι απαχθήσεις κοπέλες. Το χωριό λοιπόν αρνήθηκε να δεχθεί τα παιδιά αυτά, τα απέρριψε τα εξεδίωξε και άρα πια δεν είναι το χωριό αυτό που μεγαλώνει ένα παιδί. Σε 10, 15, 20 χρόνια πώς θα έχει μεταλλαγή αυτή η κοινωνία εξαιτίας του φαινομένου αυτού των παιδιών της Μποκοχαράμ. Σε αυτό ήθελα να σταθώ και είναι το δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησής μου. Στην εκπαίδευση. Έγινε λόγος για εκπαίδευση περί την εκπαίδευση, αλλά σκεφτούμε δύο-τρία πράγματα για τα παιδιά μας. Τον καρπό της κοιλίας μας. Όλοι αυτοί οι άντρες, οι ηγέτες, παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του Τραμπ, να, θα τον ξαναδούμε μπροστά μας. Εμείς έχουμε εξουσία και την εξουσία αυτή πρέπει να την ασκήσουμε την ώρα που τα θυλάζουμε τα παιδιά μας αυτά που θα γίνουν άντρες στο μέλλον. Να τους δείξουμε τι σημαίνει και να μην επιτρέψουμε να χαθεί αυτή η εξουσία που έχουμε ως μητέρες. Να τους μεταγγίσουμε αυτή την αξιοπρέπεια που δεν μπορούμε να έχουμε τώρα λόγω των παγκόσμιων προβλημάτων και του φόβου που επικρατεί. Φοβούμαστε τόσο γιατί κάποιοι από τους παγκόσμιους ηγέτες μιλούν κάπως διαφορετικά δεν σέβονται το, την αξιοπρέπεια της γυναίκας. Και αμέσως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διονγκώνουν την είδηση. Ναι. Μπορεί. Σε αυτό το νιερό χώρο, ένα κοινοβούλιο, να σηκωθεί κάποιος και να πει κάτι κατά των γυναικών. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό, πρέπει να το απορρίψουμε και να το στυλιτεύσουμε. Και εδώ θέλω να επιμείνω. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοιχτή, να μην αποκλεί κανέναν. Να μην παίρνει τα μάτια του άλλου για να κοιμηθεί εσύ. Να μην παίρνει τα μάτια του άλλου για να κοιμηθεί εσύ. Να κοιμάσαι με τα δικά σου τα μάτια. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε τις λύσεις κάποιων άλλων μέσα από τα δικά μας μάτια. Δεν βγαίνει όμως ο λογαριασμό αυτός. Και όταν σκεφτόμαστε για, την, ε, για στην εκπαίδευση, μπορεί σε συγκεκριμένε περιπτώσει λύσει σχετικέ με την εκπαίδευση να μην φέρουν αποτελέσματα. Γιατί μπορεί να μάθει να γράφει και να διαβάζει ένα παιδί. Αλλά να κοιτάξουμε ποιε είναι οι προσφορέ που μπορούμε να του δώσουμε, ε, ε, τι είναι αυτό που θα τα κάνει να μεγαλώσουν με γνώση, που θα του είναι όμω και οικία από την, ε, σε σχέση με την κοινωνία τους. Εγώ στην κοινωνία στην οποία μεγάλωσα, ναι, ήταν τεράστιο ε, επίτευγμα να μάθει κανείς να γράφει και να διαβάζει. Όμως μεγάλωσα σε ένα αγρόκτημα. Γελαδάρισα ήμουνα ως κορίτσι. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να προσφέρουμε στα παιδιά τη γνώση αυτή και τον πλούτο. Βεβαίως θέλουμε να δαχτούμε από τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά μην καίμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. μη χάνουμε αυτό το πλούτο και σκοιτάξουμε επικοδομητικά την εκπαίδευση, αυτή την ανοιχτή προς όλους και προς όλα εκπαίδευση πρέπει να προωθήσουμε στο μέλλον. Και εν τέλει θέλω να σχολιάσω ζητήματα για τα οποία τρέφω ιδιαίτερα έντονα συναισθήματα. Πολιτική της χειραφέτησης, της πρόσδοσης δυνατοτήτων στις γυναίκες σκλαβιά, ζητήματα αξιοπρέπειας και προσβολής της από κάποιους άλλους. Μιλήσαμε, μίλησε μία από τις ομιλήτρες για το πώς δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα, πώς δεν επιτρέπεται να μείνουμε αδρανείς. Έχουμε δύναμη, τη δύναμη την έχουμε όλες, όλοι. Μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, αλλά όλοι μαζί. Να κερδίσουμε έναν αγώνα για τη μία ημέρα, για έναν άνθρωπο, για μία χρονική στιγμή ή για μια φορά. Αλλά ας βγούμε στον δρόμο για να αισθανθούμε ποια είναι η δύναμη που φέρουμε όλοι μέσα μας. Και θα σας πω εγώ μια ιστορία τώρα για το πώς κατάφερα εγώ το δικό μου αγώνα Χωρί αυτό να σημαίνει πρέπει να τον μιμηθεί, το καθένα θα έχει το δικό του τρόπο να κερδίσει τον αγώνα του. Ξέρετε ότι έχω αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών και την αποτροπή, την κατάργηση του λιθοβολισμού ως τρόπο εκτέλεσης γυναικών υπό τον Ισλαμική Σαρία. Έχω κάνει πολλούς αγώνες, έχω γράψει δύο βιβλία. Δεν είναι όμως αυτό. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τη δύναμη των ε, παραδοσιακών ηγετών, των θρησκευτικών ηγετών και να γυρίσω εκεί από όπου ξεκίνησα. Αν έχετε διαβάσει τη βιογραφία μου θα έχετε μάθει ότι κατά λάθο ε, πήγα στο σχολείο, κατά λάθο έγινα δικηγόρο και κατά λάθο έκανα αυτόν τον αγώνα αυτό το ΣΥΠΗΝ. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω στι ρίζε μου. Ποιε είναι οι ρίζε μου όμω και ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί μου εκεί. Οι δύο καλύτεροι σύμμαχοι που έχω σε αυτή την περίπτωση είναι οι παραδοσιακοί ηγέτε και οι θρησκευτικοί ηγέτε. Έφερα λοιπόν στο Χάρβαρτ τον Σουλτάνο του Σοκουτού, γιατί είχαμε αυτή την πλατφόρμα στο Χάρβαρτ. Εκατό εκατομμύρια μουσουλμάνοι τον παρακολούθησαν. Για σταθείτε λοιπόν, τους λέει, η Σαρία δεν είναι το πρόβλημα, το Ισλάμ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι έχουν στρεβλώσει το, το Ισλάμ και την Σαρία και έχουν συνδυάσει τη Σαρία με παραδοσιακές μεθόδους. Να λοιπόν, αυτός ήρθε στο Χάρβαρτ και μίλησε. Και μάλιστα πριν μιλήσει, θέλησαμε να μας μιλήσει για ένα ζήτημα το οποίο με ανησυχεί βαθύτατα και ακόμα και σήμερα συμβαίνει, ότι δηλαδή παιδιά στην ηλικία των 10 με 12 ετών δίνονται σε γάμο σε άλλες οικογένειες. Και θέλησα να μιλήσει για το θέμα αυτό για να έχουμε τα επιχείρηματά του να τα αξιοποιήσουμε. Ήρθε λοιπόν στο Χάρβαρτ. Είχε μια μεγάλη πλατφόρμα μπροστά του. Μίλησε για την εκπαίδευση των παιδιών όπως θέλαμε και μιλώ για στρατηγικές και τακτικές. Αν ε, σκεφτείτε δηλαδή τι στρατηγικές και τακτικές σας ενδιαφέρουν εσάς, όσο μπορείτε να βρείτε από εκεί τις λύσεις. Ήρθε λοιπόν, είχαμε την πλατφόρμα όπως είπαμε του Χάρβαρτ, μίλησε. Μία από τις φράσεις που προετοιμάζοντας την ομιλία του είχαμε συμπεριλάβει ήταν ότι δεν πρέπει ένα κορίτσι να αναγκάσει να εγκαταλείψει το σχολείο για να παντρευτεί στα 8-10 του. Κάνει τη δήλωση αυτή λοιπόν δημόσια και τη φράση αυτή την πήγαμε στο χαλιφάτο, το γραφείο του δηλαδή. Και λέμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση. Την παράθεση των λόγων του. Και μου λένε ναι. Να λοιπόν σκέφτηκα, αυτή τη φράση εγώ θα την κάνω διεφημιστικό τραγουδάκι. Γιατί πιο συχνά ακούνε ράδιο οι άνθρωποι εκεί. Φροντίζαμε λοιπόν να παίζεται αυτό το τραγουδάκι Don't remove the girls out of school and marry them, άλλοι μην παίρνει τα κορίτσια από το σχολείο αλλή και για να τα παντρέψει. Το παίζαμε τι τις ωρες ακρόαση, μεγάλης ακρόασης, χρόνια αυτό το μήνυμα το διαφημιστικό και αυτή ήταν η δική μου η δυνατότητα, αυτή μου η στρατηγική, η δική μου η, η μέθοδος, εσείς μπορείτε να κάνετε περισσότερα. Και αυτό που θέλω να πω καταλήγοντα είναι ότι κανείς δεν ορίζει την αξιοπρέπειά μας, την αξιοπρέπειά μας ως γυναικών, όπως και κανείς δεν ορίζει την αξιοπρέπειά μας ως ανδρών. Μόνοι μας δεν μπορούμε, οι γυναίκες μόνοι τους δεν μπορούν, όπως και οι άντρες δεν μπορούν μόνοι τους. Τώρα που γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα των γυναικών, την Παγκόσμια μέρα των γυναικών, πρέπει να πούμε ότι όλοι μαζί πρέπει να το καταφέρουμε αυτό. Και δεν θα πρέπει να διστάσουμε να το πράξουμε. Ανεξαρτήτως της θρησκείας σας, του πιστεύω σας, του φίλου ή της σεξουαλικής σας προτίμησης, του χρώματος του δέρματός σας, να ξέρετε ότι ο καθένας σας, η καθεμία σας έχετε μια δύναμη, μια τεράστια δύναμη μέσα σας και αυτή είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτή είναι η αξία η δική σας ως ανθρώπου. Μπορείτε λοιπόν να την πάρετε στα χέρια σας και με τη δύναμη αυτή να κάνετε τον κόσμο καλύτερο για κάθε γυναίκα, για κάθε άντρα και για κάθε παιδί που ζει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τόσο πολύ για την τόσο συγκινητική αυτή μαρτυρία που μοιράστηκες μαζί μας, την προσωπική σου εμπειρία και φυσικά και το τόσο καταπληκτικό έργο σου υπερασπίζοντας γυναίκες στη χώρα σου και που τόνισε την αναγκή να αντιμετωπίσουμε την θυματοποίηση, την δημιουργία στερεοτύπων και το ότι που τόνισε ότι οι άνθρωποι, τα κορίτσια που γυρίζουν από αυτέ τι τρομερέ εμπειρίε, θυματοποιούνται και γίνονται διπλά θύματα. Και είναι απαραίτητο τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο εργασία την οικογένεια, να τους διδάσκουμε τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των γυναικών και των κοριτσιών. Θα ήθελα να αρχίσει τώρα η συζήτηση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ήδη έχουν ζητήσει το λόγο. Αν θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε ακόμα να συμπληρώσετε τα, τα έντυπα ή αν θέλετε σηκώνετε απλώς το χέρι σας για να λάβετε το. Την Αϊσέ Κεσίρ από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Παρακαλώ. Υπάρχει μετάφραση από τα τουρκικά και μην περάσετε τα δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω μέσα σε δύο λεπτά να πω όσο δυνατόν πιο σύντομα η Τουρκία είναι μια από τις πρώτες χώρες οι οποίες με το μέσο του Κοινοβουλίου του κύρωσαν τη σύμβαση των, ε, της Κωνσταντινούπολης ε, και πέρασαν το σχετική νομοθεσία με 23 άρθρα, ενώ πολλές προηγμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πλούσιες χώρες δεν έχουν ακόμη κάνει την κύρωση. Εμείς έχουμε περάσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών με 23 άρθρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα πρέπει να πω επίσης ότι η τρομοκρατική οργάνωση ΠΕΚΑΤΚΑ, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό κράτος και που ε, ε, αναγνωρίζεται και από ε, χώρες ευρωπαϊκές ως τρομοκρατική, συνεχίζει να διαπράττει τις εγκληματικές της πράξεις, να απάγει γυναίκες και παιδιά και ιδιαίτερα να άσκει βία εις βάρος γυναικών και παιδιών. Αυτά όλα έχουν δημοσιευθεί άλλωστε. Κορίτσια 15 ετών και μικρότερα με το ζόρι αναγκάζονται να πάρουν τα όπλα και να χρησιμοποιούνται ως ε, ανθρώπινη ασπίδα ή ακόμη να εκτελούνται με συνοπτικέ διαδικασίε όσοι δεν ακολουθούν. Αυτέ είναι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω. Κλείνοντα, δε, θα ήθελα να πω ότι η βία ει βάρο των γυναικών ε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την χειραφέτηση, στην πρόσδοση δυνατοτήτων και ισχύω στις γυναίκες. Βλέπουμε δυστυχώς ότι οι γυναίκες και με οικονομική ανεξαρτησία ούτως υπήν πέφτουν θύματα βίας στις χώρες φερυπίν της Ευρώπης. Εδώ χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Εξάπαντος. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Άισε είναι σημαντικό να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα από όλες τις χώρες και τις πολιτικές κατευθύνσεις για να μεταλαμπαδεύσουμε θετικές πρακτικές για να εφαρμόσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις απαραίτητες αλλαγές νομοθεσίας σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ειρήνα Σούσλιοβα από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η πρόληψη της βίας κατά των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική και στην Ουκρανία γιατί υπήρξε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία τρία χρόνια όταν ξεκίνησε η ενόπλη αντιπαράθεση στις περιοχές που ελέγχονται από το ρωσικό στρατό. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις υποχρεωτικής πορνείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και κοριτσιών. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ένοπλης σύγκρουσης υπήρξαν και μεγάλα, μεγάλη οικονομική ανεργία, ε, επιχειρήσεων, μείωση των εισοδημάτων των οικογενειών και της κοινωνικής προστασίας και αυτό οδήγησε σε μια αύξηση της εκμετάλλευσης γυναικών. Και αυξήθηκαν και οι κακομεταχειρήσεις γυναικών ακόμα και στο οικιακό χώρο. Αυτό ισχύει για όλη μας τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε κάθε κίνητρο να κυρώσουμε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατόν να αυξήσουμε <clears throat> την προστασία των γυναικών από, τις βία, από τη βία, τη βία που βασίζεται στη διαφορά του φύλου, γιατί αυτό οδηγεί σε σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά τραύματα, αλλά έχει και σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν την ισότητα των φύλων, γιατί χάρη στην ανισότητα των φύλων προκαλείται η βία. Ξέρουμε ότι η οικονομική εξάρτηση των γυναικών έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη εξάρτηση από τους άντρες και είναι πολλές φορές αβοήθητες λόγω αυτής της εξάρτησης. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Πρέπει οι γυναίκες να αποκτήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ξέρετε ότι το κοινοβούλιο μας έχει καταγγείλει την αυξανόμενη βία κατά των γυναικών στις περιοχές που είναι υπό ρωσική κατοχή και επίθεση και έχουμε και αναφορές για αυξανόμενη οικογενική βία στην περιοχή αυτή. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα η συνεδρίαση Μικτή Επιτροπή με το Ουκρανικό Κοινοβούλιο και εγώ θα ήθελα πράγματι στα πλαίσια αυτά να θίξω αυτό το θέμα και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να προωθήσουμε την κύρωση τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. Το λόγο στη συνάδελφό μου το Ελληνικό Κοινοβούλιο Αφροδίτη Σταμπόγλη, που είναι η πρόεδρο τη Επιτροπή Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα των Φίλων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τις ομιλήτριες για τις ε, τοποθετήσεις τους. Θα ήθελα να πω ότι η βία κατά των γυναικών και η καταπολέμησή της είναι θέμα που αναδείχθηκε από το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας. Σταθμό στην αντιμετώπιση του φαινομένου αποτέλεσε η ψήφιση του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία το 2006, ο οποίος προβλέπει αυτεπάγγελτη δίωξη των δραστών, προστασία των θυμάτων και ποινικοποίηση στο βιασμό μέσα στο γάμο. Ακολούθησε η ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία Οδηγιών για τη Σεξουαλική Παρενόχληση στον χώρο της εργασίας, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, που όπω ξέρουμε αφορά κατά 80% γυναίκες και κορίτσια και επίσης η κύρωση της Σύμβασης της Βαρσοβίας ε, και η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την υποστήριξη των θυμάτων τράφικινγκ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κύρωση της οποίας συστάθηκε αυτές τις μέρες νομοπαρασκευαστική επιτροπή και η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει τις πραγματικές προϋποθέσεις ώστε η κύρωση να μην παραμείνει ε, γράμμα κενό. Από το 2011 άρχισε να υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας η λειτουργία 39 συμβουλευτικών κέντρων και 21 κέντρων φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας. Την ίδια χρονιά άρχισε να λειτουργεί η συμβουλευτική γραμμή ΣΟΝ στα ελληνικά και στα αγγλικά 24 ώρες το 24ωρο και από τη σύνθεση των γυναικών που απευθύνθηκαν ε, για συμβουλευτική και υποστήριξη διαπιστώνουμε ότι 27% από αυτές ήταν εργαζόμενες και οι μισές αυτοπασχολούμενες, 15% είχαν μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και 10% δήλωσαν ότι είχαν καλή ή πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Άρα συμπεραίνουμε ότι όσο αναγκαία είναι η υποστήριξη της οικονομικής ανεξαρτητοποίησης των γυναικών ώστε να μην ανέχονται τη βία σε βάρος τους, άλλο τόσο είναι αναγκαία η αμφισβήτηση των πατριαρχικών στερεοτύπων μέσα στην κοινωνία. Το γεγονός επίσης ότι μόνο 8% δήλωσαν μετανάστριες, 1% άτομα με αναπηρία και 1% μέλη μειονότητας τεκμηριώνει ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες απευθύνονται δυσκολότερα ή δεν έχουν καν πρόσβαση στη συμβουλευτική και την υποστήριξη. Σε αυτές τις πιο ευάλωτες ομάδες λοιπόν απευθύνεται τώρα πια η Γενική Γραμματεία, ιδιαίτερα η Γενική ε, Γραμματεία Ισότητας έχει προβεί σε εμπλουτισμό της λειτουργίας των συμβουλευτικών κέντρων με συμβουλευτική εργασία ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους, γίνονται καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημερωτικό υλικό σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά και τουρκικά στην περιοχή όπου κατοικεί η μουσουλμανική μειονότητα τουρκόφωνη στην ε, πλειοψηφία της. Υπάρχουν μηνύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο μεταναστευτικό τύπο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιστοσελίδα και facebook. Με τη βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπαιδεύονται σύμβουλοι, νομικοί υποστηρικτές, αστυνομικοί, υγειονομικοί και δικαστικοί, ώστε να προσανατολίζονται σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Από το Τώρα, όσο ε, επίσης αυτά τα κέντρα μετά την εμφάνιση του προσφυγικού κύματος το 2015 ε, δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που θεωρούνται θύματα βίας και μέχρι στιγμής έχουν ε, φιλοξενήσει ένα διψήφιο αριθμό γυναικών προσφύγων με τα παιδιά τους. Ε, συνιστάται στους υπεύθυνους ε, των ε, camps όπου διαμένουν πρόσφυγες και των επιτροπών... Παρακαλώ, είναι μεγάλος ο κατάλογος των αγορητών, λυπάμαι. 30 ε, δευτερόλεπτα. Ε, συνιστάται στους υπεύθυνους των Επιτροπών Ασύλου η εντόπιση θυμάτων βίας και θυμάτων τράφικινγκ ή θυμάτων σε κίνδυνο για πρόημο γυναικών σε κίνδυνο για πρόημο καταναγκαστικό γάμο ή ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένα για το πόσες γυναίκες έχουν πάρει άσυλο για τέτοιους λόγους, για το πόσο σωστά τηρούνται αυτές οι οδηγίες. Ευχαριστώ για την ανοχή σας very much, Ευχαριστώ πολύ, Αφροδίτη. Λυπάμαι, τη συνάδελφοι. Πρέπει να παραμείνουμε μέσα στο χρονικό μας πλαίσιο, γιατί συνέχεια μου ζητούν να λάβουν το λόγο και θέλω να δώσω το λόγο σε όλους αυτού που θέλουν να συμβάλλουν. Θέλω να σου πω, Αφροδίτη, όμως, ότι είχαμε μια επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή των Γυναικών που πήγε στην Ελλάδα και εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα με το καταφύγιο αυτό γυναικών, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε πόσο καλή εργασία έχει κάνει και σε άλλες χώρες έχουμε επισκεφθεί και καταβλισμούς προσφύγων όπου υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα για την ασφάλεια των γυναικών και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα και ιδίως αυτό για την μεταρρύθμιση του πακέτου ασύλου έχουμε ζητήσει να υπάρχουν χωριστές υγειονομικές εγκαταστάσεις για τις γυναίκες και περισσότερη ασφάλεια και παρουσία αστυνομία στη νύχτα. δυστυχώ, στα, στους καταβλισμούς προσφύγων υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες που την χάνουν θύματα παρενόχλησης. Τώρα δίνω το λόγο στη, στη Λέτα Ντελίν από το Κωσυφοπαίδιο που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών του Κοινοβουλίου του Κωσυφοπαιδίου. Open the mic, please. Ανοίξτε το μικρόφωνο, παρακαλώ. Θα μιλήσω αλβανικά αν γίνεται. Υπάρχει μετάφραση πιστεύω. I'm sorry we don't have Albanian. Έχουμε. Δεν έχουμε αλβανικά λέει πρόεδρος. Yes, yes, we have, transla we have a translation in Albanian. Uh, thank you. Faleminderit. Uh, uh, Përshëndes të krejt Σας ευχαριστώ και χαιρετίζω όλους τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπατε προηγουμένως, εκπροσωπώ την, ε, τους γυναίκες βουλευτές στο Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου. Έχω παρακολουθήσει με συγκίνηση τις προσωπικές εμπειρίες των ομιλητριών και νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να είμαι εδώ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Νομίζω και οι συναδελφοί μου συμμερίζονται αυτές τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες και αποστασιοποιούνται πλήρως από τις βίες ενέργειες και τα επιθετικά λόγια τα οποία ακούστηκαν σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να αναφέρω και ένα θέμα που αναφέρθηκε και εδώ προηγουμένως. Υπάρχουν 20.000 γυναίκες από το Κωσυφοπέδιο που έπεσαν θύματα βιασμών από Σέρβους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάποιες από αυτές έχουν καταφέρει να επανασωματωθούν στην ε, κοινωνία όπου ζούσαν στην τοπική κοινωνία του πεδίου και έχουμε πρόσφατα περάσει νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κατοποίησης σε καιρό πολέμου. Πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η πιο πρόσφατη έκθεση για το ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να αναφέρω ότι κάποιοι στρατιωτικοί στρατηγοί από την πλευρά της Σερβίας έδωσαν εντολή συστηματικού βιασμού των γυναικών του Κωσυφοπεδίου και τώρα παρασημοφορούνται στην δημοκρατία της Σερβίας. Εμείς καταδικάσουμε αυτές τις ενέργειες και οι γυναίκες αυτές που έτυχαν βιασμού κατά τη διάρκεια του πολέμου διεκδικούν δικαιοσύνη. Και αυτή η δικαιοσύνη τους, τους έχει αρνηθεί η Σερβία. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή της ε, Παγκόσμιας της γυναίκας, ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει δικαιοσύνη για όλες τις γυναίκες, μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες του κοσφοπεδίου. Τα θέματα αυτά τα έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους μας από τη Σερβία. Ζητάμε να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτές που δεν έχουν πετύχει αυτή την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πρέπει να γίνει με την πίεση και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που δεν είναι ακόμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να καταδικάσουν αυτές τις αποτρόπιες ενέργειες που είναι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρος. Ήμουνα για έξι χρόνια παρούσα στους πολέμους των Βαλκανίων. Κατανοώ πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε και η αντιμετώπιση της αντιμορρησίας από όπου και αν προέρχονται τα εγκλήματα κατά των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Η χρήση του βιασμού ως όπλου στον πόλεμο, αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να λαμβάνει η χώρα σε πάρα πολλά μέλη του κόσμου και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Και τώρα, συνάδελφος από την Ισπανία, η Νάγια Αλμπακοβέλη από την Επιτροπή για την Ισότητα. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις ομιλήτριάς μας για το θάρρος τους και τη συγκινητική μαρτυρία που κατέθεσαν εδώ. Τα στοιχεία που έχουμε από την Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες σε ό,τι αφορά τους θανάτους από την σεξιστική βία είναι πραγματικά ανασυχητικά. Έχουμε γυναίκες, πολλές γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί και υπάρχουν και περιπτώσεις ακόμα που είναι υπό έρευνα. Όλα αυτά συνδέονται ιδιαίτερα με αυτά που είπαμε στην αρχή για το θέμα της οικονομικής ανέχειας. Έχουμε 24% μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολλές γυναίκες οι οποίες είχαν την οικονομική τους ανεξαρτησία, <clears throat> αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν στους ε, ε, πρώην συζύγους τους και αυτό έχει αυξήσει την οικονομική, την ε, βία που υφίστανται αυτές οι γυναίκες, οι οποίες τώρα εξαρτώνται από τους συντρόφους τους για να επιβιώσουν και φυσικά δεν τολμούν να καταγγείλουν αυτή τη βία που υφίστανται στο σπίτι. Ποτέ λοιπόν δεν έχουν καταγγείλει πολλές από αυτές γιατί υπάρχει το πρόβλημα της οικονομικής τους ε, εξάρτησης από αυτόν που τους κακοποιεί. Και αυτές οι οικονομικές διαφορές που έχουν οξυνθεί λόγω της κρίσης που δεν δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να κερδίσουν το ψωμί τους όταν μεγαλώσουν δεν έχουν συμπληρώσει αρκετές μέρες εργασίας για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και υπάρχει και βία εναντίον των πιο ηλικιωμένων γυναικών. Έχουμε λοιπόν ένα μακρύ δρόμο να διατρέξουμε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις δολοφονίες στη δική μας περίπτωση στα ισπανικά κόρτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εργασία μιας υποεπιτροπής που αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα κέρια θέματα τα οποία είναι σημαντικά για όλες Είναι και στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Νάντια. Απλώς να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή ακριβώ έχουμε μια έκθεση που εξετάζεται στο Κοινοβούλιο για το μισθολογικό χάσμα ε, και για το χάσμα στι συντάξει. Πέρασε η πρώτη την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Συνάδελφοι, θα πρέπει δυστυχώ να κόψω τι παρεμβάσει σα στο ένα λεπτό, διότι έχουμε τόσε πολλέ ε, ε, αιτήσει για να λάβουν το λόγο οι συνάδελφο. Η Μάθα τώρα από το Κοινοβούλιο του Μαρόκο. επί σειρά ετών η καταπίεση εις βάρος των γυναικών βασιζόταν σε επιχειρήματα θρησκευτικού χαρακτήρα. Στο όνομα του Θεού και του Ισλάμ εξανδραπονδίζονταν και τους αποστερούσαν κάθε τους δικαίωμα. Ωστόσο, χωρίς να ξεκινήσουμε μια συζήτηση θεολογικού χαρακτήρα, θα αρκούσε να δούμε τις απαρχές του Ισλάμ για να εντοπίσουμε τα λαμπρά παραδείγματα γυναικών που είχαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική της εποχής. Η γυναίκα του προφήτη, η Χαντιζά, που παντρεύτηκε τον προφήτη και αυτό δεν την εμπόδισε να συνεχίσει το εμπόριο. Η γυναίκα του, η Χαΐσα, όπως είχε διευκρινίσει και ο προφήτης, έπρεπε να σπαστεί τη θρησκεία μεν, αλλά είχε την δική της συμβολή μαζί με τις υπόλοιπες ε, γυναίκες που συμμετείχαν στο ανώτατο συμβούλιο, το συμβούλιο που λάμβανε τις ε, σημαντικότερες κρατικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ουαφ. Και τώρα η Τζούλι Γουόρντ, συναδελφός μου, η οποία ε, συμμετέχει μαζί μου στην ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καθήκον να είμαστε ιδιαίτερα αυστηρές για τόσο συμβαίνουν στις δικές μας τις χώρες. Εδώ πρέπει να υψώσουμε τον αστιμά μας και να στηρίξουμε πολιτικές στρατιωτικές δυνάμεις ή υπουργού να υποστηρίξουμε την καταδίκη αξιωματούχων, υπουργών, στρατιωτών που έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά των γυναικών. Και στη δική μου τη χώρα πρέπει να ε, ασκηθεί πίεση για να κυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσω την κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία. Από ό,τι ξέρω, στα σύνορα με το Κορδιστάν υπάρχει εκεί συνενοχή μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και κάποιων τζιχαντιστών που πιέζουν τις γυναίκες και τις οδηγούν στην, στην αγοραπολισία ως ε, σεξουαλικών σκλάβων. Όλες μας οι κυβερνήσεις, όλοι μας οι, υπουργού, οι υπουργοί πρέπει να αναλάβουν αμέσως δράση για την πρόσπιση αυτών των γυναικών που είναι πλέον ευάλωτες. Υπάρχουν ακόμη και αποδείξεις, τιμολόγια, αποδείξεις από τις αγοραπολισίες των γυναικών σε αυτά τα κείμενα. 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια φτάνει ο τζίρος αυτού του εμπορίου. Είναι απίστευτο. Πρέπει να ασκήσουμε κριτική κατά των δικών μας των κυβερνήσεων. Υπάρχουν γυναίκες στην Τουρκία που είναι κλεγμένες στην Τουρκία ε, νομίμως και είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να καθόμαστε να λέμε τι ωραίο είναι να υπογράφει κανεί μια χάρτα και να προσχωρήσει μια σύμβαση ενώ υπάρχουν γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή, τα σώματά τους ε, πολλούνται και αγοράζονται και είναι θύματα εμπορίου, διακίνησης. Σε ευχαριστούμε Τζούλη. Σε ευχαριστούμε Τζούλη. Ε, διαρκώς υψώνουμε τη φωνή μας, καταδικάζοντας την κατάσταση στην Τουρκία και για τους φυλακισμούς και το ΠΚΚ που θεωρείται ως τρομοκρατική οργάνωση Μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε αυτόν τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας λοιπόν σε όλα τα μέτωπα κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Η Λένα Γιάννησεν από τη Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω μερικά λόγια. Για ορισμένες αναφορές σχετικές με τη βία που όλο και περισσότερο επικρατεί στις κοινωνίες μας. Βία που βλέπουμε στο Μάλι αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Εμείς στο κοινοβούλιο μας είδαμε μια έκθεση για τις γυναίκες θύματα βίας ένοπλων συγκρούσεων και είναι σημαντικό αυτό να το δούμε και να φέρουμε το θέμα στο υψηλότερο επίπεδο συζήτησης και στο δημόσιο διάλογο. Μάλιστα διάβασα και την ε, τελευταία πρόταση νόμου στη Ρωσία, αυτή που πέρασε μειώνοντας την ποινή εις βάρος ανδρών που καταδικάζονται για κακοποίηση των συζύγων τους. Εμείς στην Σουηδία έχουμε ακριβώς την αντίστροφη τάση, δηλαδή ο νόμος ο οποίος αφορά τον βιασμό πλέον ρητά αναφέρει πως βιασμός υπάρχει μέσα στην οικογένεια, είναι καταδικαστέος, δεν επιτρέπεται ο σύζυγος να βιάζει την σύζυγο και αυτό οδηγεί σε καταδίκη ε, σε ποινή φυλάκιση μεγαλύτερη όταν έχει βιάσει τη σύζυγό του. Και είναι πολύ σημαντικό να αγωνιστούμε για αυτά τα προβλήματα στις διάφορες χώρες και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε σου ειδικά η Πρόεδρος. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε και σε αυτή την νομοθεσία, το νέο νόμο από την ε, Δούμα της Ρωσίας, η οποία ουσιαστικά αποποινικοποιεί τη βία εις βάρος των γυναικών. Άπαξ και η βία αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στην οικογένεια. Και μάλιστα ποινικοποιεί και τη βία βάρο των παιδιών. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήμασταν πολλοί βουλευτέ που ψώσαμε τη φωνή για να εκδηλώσουμε την ελεγγύη μα προ τι γυναίκε αυτέ που πέφτουν θύματα βία ενδοοικογενειακή στη Ρωσία. Δίνω το λόγο τώρα στην ε, ε, Ράφια Ελμασούση από το Κοινοβούλιο του Μαρόκου. Ε, Καλημέρα σας. Ραφιαέλ Μανσουρί. Ε, άκουσα τις ε, ομιλίες νωρίτερα, τις εμπειρίες από τις διάφορες χώρες που αναφέρθηκαν και θα ήθελα και εγώ ε, ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου μου, ως γυναίκα μαροκινή να σας μιλήσω για τα επιτεύγματα της χώρας μου στην τελευταία δεκαετία. Όπως γνωρίζετε είναι αναπτυσσόμενη χώρα του Μαρόκο. Υιοθετήσαμε λοιπόν το 2011 νέο σύνταγμα, στο οποίο εισάγεται η αρχή της, ε, καθιερώνεται μάλλον η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ας μιλήσουμε λησμονούμε ότι ο οικογενειακός κώδικας δίνει δικαιώματα στη γυναίκα ως ε, σύζυγο και μητέρα. Έγιναν πολλοί αγώνες για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, κυρίως γυναικών και κοριτσιών στις περιοχές της Υπέθρου. Αναπτύχθηκαν προσπάθειες για την προαγωγή των γυναικών στις περιοχές αυτές και προσπαθούμε και να ενισχύσουμε την ε, κοινωνία των πολιτών με περισσότερη ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της. Βεβαίω ε, διαπράττονται πράξεις βία ει βάρο των γυναικών, αλλά όσον αφορά τη βία, την ενδοοικογενειακή και αυτό που ανέφεραν οι προηγούμενε ομιλήτριε θα ήθελα να πω ότι ελπίζουμε όλοι να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Um, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Ράφια. Η κυρία Χάνιμαν, αγαπητή συνάδελφος. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε όλοι. Μιλούμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό και ήθελα να θέσω το ζήτημα της καταγγελίας της ενδοοικογενειακής βίας και των ενδο οικογενειακών βιασμών. Γιατί πολλές φορές μας έχουν απασχολήσει τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το οικογενειακή βία και ο βιασμός από το σύζυγο, αλλά πολλές φορές διστάζουν οι γυναίκες να, κατα... να καταγγείλουν και βέβαια και ο αριθμός των ε, καταδικών φαίνεται μάλλον να παρουσιάζει μειωτική τάση. Δεν νομίζω ότι έχουν μειωθεί οι βιασμοί μες στο γάμο. Μάλλον για κάποιους λόγους οι γυναίκες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις αρχές, στις νομικές αρχές και αυτό είναι ένα πρόβλημα βεβαίως γιατί εάν δεν μπορέσουμε στις χώρες μας να φτάσουμε σε μια θέση όπου οι γυναίκες θα αισθάνονται κάποια εμπιστοσύνη στις αρχές επιβολής της τάξης και του νόμου δεν είναι δυνατό να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, τουλάχιστον όχι κατά τρόπο ικανοποιητικό και καλό όσο θα θέλαμε. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν και το άλλο, το ζήτημα το σχετικό με την πορνεία, γιατί έγινε λόγος βέβαια για την ε, διακίνηση ανθρώπων ε, η οποία τροφοδοτεί την ε, πορνεία. 85% των εργαζομένων στην πορνεία για σεξουαλική εκμετάλλευση, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Στατιστικές έχει περάσει από τα λαθρέα δίκτυα διακίνηση ανθρώπων. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί και νωρίτερα τώρα το απόγευμα, μια συνεδρίαση μιλούσε για το σκανδιναβικό του σοπίν μοντέλο, όπου αυτός ο οποίος ε, παίρνει, δέχεται τις σεξουαλικές υπηρεσίες είναι ο ένοχος και όχι η πόρνη. Αντίστροφα δηλαδή από αυτό που ισχύει στο γερμανικό και γενικά υπηρετικό σύστημα. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σαν λύση, δηλαδή πάντα να βλέπουμε ως ένοχο εκείνον ο οποίος προσφεύγει στις υπηρεσίες τις σεξουαλικές. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην άλλη συνάδελφα από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, την Σαντεμίρ Τσελίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έρχομαι από, μια, από ένα κοινοβούλιο ηρωικό, την ηρωική τουρκική εθνοσυλλήψη, έτσι λέγεται στα τουρκικά, και από μια ηρωική πόλη, το Αντεπ, το ηρωικό Άντεπ. Είμαστε λοιπόν μια συνέλευση ηρωική, η οποία μπόρεσε να αντισταθεί και σε ένα φωνικό πραξικόπημα που κόστησε τη ζωή 11 γυναικών που αντιστάθηκαν σε αυτό τον Ιούλιο του 2016. Προέρχομαι, όπως είπα, από το ηρωικό Αντέπ, από τον Καζή Αντέπ. Σήμερα, με την ημέρα των γυναικών, θα ήθελα να τιμήσω τις γυναίκες που ε, λόγω της μεγάλης κρίσης στη Συρία έχουν πέσει θύματα ε, βίας. Ύστερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Συριακή κρίση είναι εκείνη η οποία έχει κοστίσει τα περισσότερα θύματα. Το 2011 είχαμε 250, ε, περάσματα καθημερινά, ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη χώρα μου από τη Συρία. Είναι τεράστιο λοιπόν το προσφυγικό ρεύμα και το ΑΝΤΕΠ είναι μια από τις χώρες οι οποίες έχει υποστεί ε, τις μεγαλύτερες ε, πιέσεις ε, πάνω από 150.000 50.000 ανθρώπους έχει υποδεχθεί το Αντέπ ε, ως πρόσφυγες και πολλοί από αυτούς, μεγάλο από αυτούς, ζουν μέσα στην πόλη. 1,4 εκατομμύρια είναι τα παιδιά από τη Συρία που υποδεχόμαστε. Από τα 3 αυτά εκατομμύρια, 1,3 εκατομμύρια είναι γυναίκες πρόσφυγες. Με πολύ μεγάλη ευαισθησία και αυτοθυσία τους υποδεχόμαστε και τους προσφέρουμε, γιατί η μόνη μας προσέγγιση είναι η ανθρωπιστική προσέγγιση. Ανοίξαμε τις φύλες, προσφέραμε ε, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματική αποκατάσταση, κάθε είδους υπηρεσία και ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες δίνουμε προτίμηση με το σύστημα των θετικών προτιμήσεων. Ιδιαίτερα στα θέματα της προσωπικής υγιεινής δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών οι γυναίκες και τα παιδιά. Όπως και οι άλλες ευάλωτες ε, ομάδες έχουν στη διάθεσή τους και προσωπικό ασφαλείας, 1500 κάμερες ασφαλείας και όσο το δυνατόν πιο αυστηρή φύλαξη και ιδιαίτερες συνθήκες για τις γυναίκες της εγγύους και τις θυλάζουσες. Σε αυτές διαθέτουμε επί παραδείγματι στην ε, φυλάδια ενημερωτικά στην αραβική γλώσσα. Ε, προσφέρουμε μαθήματα, ε, μιλούμε για την βία εις βαρός των γυναικών, για την ισότητα και απευθυνόμαστε στην κατάλληλη γλώσσα στις γυναίκες αυτές. Πολλές συνεδριάσεις έχουμε οργανώσει, έχουμε προγράμματα οικογενειακού εκπαίδευσης, έχουμε εκπαιδεύσει δασκάλους, δασκάλες ε, και προσφέρουμε διδασκαλία και μαθήματα στις γυναίκες από τη Συρία. Και πρέπει, αγαπητοί, φίλοι, σας ε, παρακαλώ ειλικρινά να τελειώσετε την ομιλία σας. Έχετε βεβαίως ένα πολύ σημαντικό θέμα να εκθέσετε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρονικό περιθώριο. Σας ευχαριστώ. Λέει η κυρία με συγχωρείτε που σας διακόψα, είναι τόσο σημαντικά αυτά που είπατε και μάλιστα έχουμε επισκεφθεί το Γκαζιαντέπ με επίσημη την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συναντήσαμε την δήμαρχό σας. Ξέρουμε πολύ καλά τα όσα γίνονται στο ΑΝΤΕΠ και δεν θέλω καθόλου να μειώσω την προσφορά σας. Αυτά τα οποία πράτετε αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη και δεν ήθελα να υπονομέσω την ε, τοποθέτηση σας. Αλλά έχουμε τελευταία ομιλήτρια την κυρία Πάολα Μπρέμερ από την Σουηδική Βουλή. Ευχαριστώ. Είμαι η εισηγήτρια και σε άλλο σεμινάριο και πρέπει να βιαστώ. Δεν θέλω να συμμετάσχω ακριβώς στην ε, συζήτηση, διότι αισθάνομαι ευλογημένη στη Σουηδία. Είμαστε προφυλαγμένοι από όλα τα προβλήματα που ακούσαμε να παρουσιάζονται. Όμως έχω μια ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις γυναίκες που είναι εχμάλωτες του ΝΤΑΕΣ. και με τους θρησκευτικού ηγέτες. Τι συνεργασία μπορούμε να έχουμε στη Σουηδία. Το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε είναι να έχουμε μια κοινωνία διχασμένη στο επίπεδο των ε, θρησκευόμενων. Και όσοι είναι πνευματικοί τάγοι, δυστυχώ είναι περισσότερο υπεύθυνοι για ριζοσπαστικότερα κινήματα. Δεν εκπροσωπούν του καθημερινού μουσουλμάνου τη Σουηδία, για να το πω έτσι. Έχετε καμιά ιδέα τι να κάνουμε, τι να κάνουμε για να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι λάθος ηγέτες. Σε ευχαριστώ, Παόλα. Για να ολοκληρώσουμε, ο λόγος στην ε, Λάμια και την Χάουα για δύο τελευταίες κουβέντες. Και εσείς θα έχετε τον λόγο αύριο. Λυπούμε, δεν έχουμε χρόνο. Είχαμε ε, δημοσιεύσει μια κοινή δήλωση, κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων, Επιτροπή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο Προεδρεύουσα χώρα, ε, που ε, ε, προέκυψε από την διάσκεψη της Μάλτας, Μάλτα η οποία τώρα έχει την Προεδρία, Εκεί είναι η δήλωση. Βλέπετε πώ προσπαθούμε να ενώσουμε τι δυνάμει των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να υπάρξει μηδενική ανοχή στην ατιμορρησία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λάμια, χάουα. Εντάξει, κινήστε εσεί ανάποδα. Περνάει ο χρόνο. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Μονάχα το γεγονό ότι μπορώ να ακούσω τι απόψει εκπροσώπων από διαφορετικέ χώρε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το θαυμάσιο, το εκπληκτικό. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για όλε μα. Αλλά να πω μονάχα αυτό και θα στριοποιήσω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω. Έχουμε πολλές συζητήσεις για τους πόρους. Θα πρέπει να Έχουμε πολλούς πόρους, αλλά αν η γυναίκα δεν έχει πρόσβαση στους πόρους αυτούς, δεν ωφελούν σε τίποτα. Η πρόσβαση στους πόρους, η λογοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεύτερον, πρέπει να ξανασκεφτούμε γιατί είμαστε εδώ. Τι κάνουμε εδώ. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα πάνελ, περισσότερες συζητήσεις, μα δεν έχουμε συζητήσει αρκετά πια γιατί είμαστε εδώ και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι τόσο πολλά αυτά που θέλουμε να κάνουμε και ας το κάνουμε σε επίπεδο πράξης. Όχι απλώς να μιλάμε, αλλά να δράσουμε. Και τέλος, το μυαλό μας και η καρδιά μας θα πρέπει να είναι στο σωστό μέρος. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον δικό μας προσωπικό χώρο, στο δικό μας περιβάλλον η κάθε θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά ας ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο κόσμο για τις επερχόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Και η Λάμια τώρα για τις τελικές παρατηρήσεις. ο καθένας από εμά, η καθεμία από εμά θα πρέπει να εργαστεί, να καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες που είναι ακόμα στα χέρια του Ντάες, του Ισλαμικού κράτους. Όλοι ξέρουν ε, πόσο έχουν υποφέρει αυτές οι γυναίκες και τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Υπάρχουν γυναίκες και παιδιά στα χέρια του Ντάες που ε, βιάζονται και παιδιά ακόμα που είναι μικρότερα από 8 χρονών. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε για να σταματήσει πια αυτό. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να κλείσω με αυτήν την με αυτή την ε, έκκληση για δράση. Χειροκροτήστε παρακαλώ και δώστε έτσι την υποστήριξή μας. Και ευχαριστώ για αυτή την τόσο πλούσια συζήτηση και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενωμένοι βοηθώ, με τη βοήθεια και των κρατών μελών για να υπάρξει η κύρωση τουλάχιστον στην Ευρώπη της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστώ. Και τώρα μια οργανωτική ανακοίνωση. Ναι, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Για αυτούς που θα είναι στο εργαστήριο υπαριθμό 5 για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και τους στόχους της ε, ε των Εθνών Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ξεκινήσει τώρα αυτό το εργαστήριο. Όσοι, όσες πάνε στο εργαστήριο 4, ισότητα ανδρών και γυναικών, πάτε στην αίθουσα PHS 1002 θα σας ε, οδηγήσει εκεί ένα μέλος της γραμματείας και ελπίζω ότι θα είστε όλοι παρούσες στις 6.45 για την τελετή που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ.